I would like to start the meeting because we are... Να ξεκινήσουμε. Καλημέρα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. I would like to welcome eh, everybody. Να καλωσορίσω όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ, τόσο νωρίς. Θέμα στην συνταγματική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συζητήσουμε σήμερα το ζήτημα των δικαιωμάτων των πολιτών και για το σκοπό αυτό έχουμε ζητήσει από το Τμήμα Πολιτικής να εκπονήσει μία έκθεση, μία μελέτη. Θα μας την παρουσιάσουν οι δύο καθηγητές που ήταν επικεφαλής της ομάδας που εκπώνησε την μελέτη αυτή. Δεν είναι ακόμα έτοιμη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε μια εβδομάδα θα γίνει αυτό, αλλά σήμερα θα ακούσουμε τους δύο καθηγητές. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή... Ah, no translation. Α, δεν υπάρχει ακόμα διερμηνία, λέει η Πρόεδρος. I see English. Uh, Βλέπω όμως ότι η διερμηνής είναι εδώ. Επομένω, κανονικά θα έπρεπε να λειτουργεί. Βρείτε το κανάλι σας παρακαλώ. Uh, Έχουμε λοιπόν δύο καθηγητές οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν αυτή τη μελέτη. Είναι ο καθηγητής Αντώνιο Φερνάντες Τομάς και, και ο καθηγητής Διέγο Λόπες Γκαρίντο από το Πανεπιστήμιο Καστίγια Λαμάντσα Ένας είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου και ο άλλος είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Θα ακούσουμε δηλαδή και δύο διαφορετικές οπτικές. Το δυστύχημα σήμερα είναι ότι έχουμε μια πολύ σοβαρή ψηφοφορία για μια πολύ δύσκολη έκθεση. Είναι πάρα πολύ ε, μεγάλη σε διάρκεια θα είναι αυτή η ψηφοφορία και στις 11.30 θα πρέπει να τελειώσουμε την ε, συνεδρίασή μας για να πάμε στον ε, πανηγυρικό εορτασμό του Κοινοβουλίου για την επέτειο των 60 χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, οπότε δεν μπορούμε να, να ξεπεράσουμε τον χρόνο που έχουμε προβλέψει, δηλαδή μέχρι τις 10. Θα δώσω λοιπόν κατευθείαν τον λόγο στους καθηγητές για να μας κάνουν την παρουσίαση. Θα γίνει συζήτηση μέχρι τις 10. Θα συζητήσουμε λοιπόν τα ζητήματα που σχετίζονται με το Brexit τα επόμενα δύο χρόνια. Φυσικά θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και στην πορεία του χρόνου τα επόμενα δύο χρόνια. Ο κύριος Αντώνιο Φερνάντες Τομάς έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας ε, δια την ε, τιμή που κάνετε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό των Ευρωπαίων πολιτών και είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας μαζί με τον συνάδελφό μου Διέγκο Γκαρίδο για να σας ε, μιλήσω για το θέμα αυτό. Λέγομαι Αντώνιο Φερνάντο Τομάς και είμαι καθηγητής διεθνούς ε, και ε, δημοσίου δικαίου στην Καστilla Λαμάντσα. Θα σας αναφερθώ, θα σε έξι στοιχεία του πρώτου τμήματος της έκθεσης σχετικά με το Brexit και των κεκτημένων δικαιωμάτων της των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχα αντίστροφα. Φοβούμαι ότι δεν είχατε και πολύ χρόνο έτσι ώστε να εξετάσετε την πρώτη εκδοχή της έκθεσης και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι εγώ έχω συγγράψει το πρώτο τμήμα, όπως άλλωστε το είπε ε, και η κυρία Πρόεδρος ε, και ο συνάδελφός μου ασχολήθηκε με το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντα υπόψη τα στοιχεία αυτά λοιπόν, θεωρώ σημαντικό ε, να σας πω ότι τα εννέα συμπεράσματα τα οποία σχετίζονται με το πρώτο τμήμα δεν βρίσκονται στο τέλος αλλά ανάμεσα στη σελίδα 30 και 33 του εγγράφου. Τα συμπεράσματα λοιπόν έχουν, ε, αριθ, έχουν ε, συγκεκριμένη αρρύθμιση ε, και έχουν συγγραφεί με τρόπο σαφή έτσι ώστε να γίνει αμέσως κατανοητό το περιεχόμενό τους. Εγώ θα ασχοληθώ τώρα με τα έξι στοιχεία της σύνοψης. Πρώτον, θεωρώ σκόπιμο να ξεκινήσω λέγοντας ποια είναι τα κεκτημένα δικαιώματα. Πρόκειται για υποκειμενικά δικαιώματα των πολιτών, τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε ένα νομικό <clears throat> συγκεκριμένο πλαίσιο και ε, ε, με οποιαδήποτε, παρά οποιαδήποτε αλλαγή στην ισχύουσα νομοθεσία, ε, εξακολουθούν να ισχύουν και σε άλλο διαφορετικό από το αρχικό νομικό σύστημα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ε, έδωσαν, έδωσαν ε, δικαιώματα ε, κατάσχεσης από πλευράς των κρατών με αξίωση αποζημίωσης των πολιτών που είχαν φυγεί. Το 1917 δύο ψηφίσματα ε, των ε, δύο βουλών ε, του Ηνωμένου Βασιλείου έδωσαν μια νέα τροπή σε αυτά τα κεκτημένα δικαιώματα και για προστασία των ε, πολιτών ε, της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από την απόσταση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αυτό σε περίπτωση που θα υπάρξει λοιπόν τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος που δεν θα είναι πλέον για αυτούς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά το δίκαιο της κάθε χώρας μέλους την οποία θα ζουν. Πρέπει πάντως να μην λησμονούμε ότι υπάρχει ε, πάντα η άγνωστη παράμετρος, ε, δηλαδή εάν είναι δυνατόν να δοθούν σε ένα πλαίσιο διαφορετικό από το αρχικό, αλλά επίσης και ε, ε, ε, σε προάσπιση άλλων δικαιωμάτων που δεν αφορούν την ιδιωτική περιουσία, αλλά θα αφορούν, ας πούμε, βασικές προσωπικές ελευθερίες ή τα όσα περιλαμβάνονται στο καταστατικό των Ευρωπαίων πολιτών. το, ε, ε, πρέπει να υπάρξει κάποια διασύνδεση ανάμεσα ε, στα στοιχεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Δεύτερο. Είναι δυνατόν να εξευρεθεί συγκεκριμένο συμπέρασμα διαβάζοντας την ομολογία σχετικά με την έννοια των κεκτημένων ε, δικαιωμάτων που δεν έχουν ε, εφαρμοστεί στις ε, βασικές εμπορικές ε, ε, έννοιες όπως ας πούμε δικαίωμα εγκατάστασης, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ. Όσον αφορά ε, το ιδιωτικό, την ιδιωτική κτήση υπάρχουν ήδη κάποια παραδείγματα στην Άνω τα δικαιώματα της Γερμανίας ή στην Πολωνία. Η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει την ύπαρξη μιας γενικής αρχής σεβασμού των κεκτημένων δικαιωμάτων των ιδιωτών. Ωστόσο, αυτή η αρχή, εάν τότε όντως ίσχυε, παρόλα αυτά ε, είχε ε, και περιείχε ε, κάποιες εξαιρέσεις βάσει της σύμβασης της Γενέβης που τότε αποτελούσε την νομική βάση <clears throat> στην διάρκεια της αντιδικίας σε σχέση με το ισχύον πολωνικό δίκαιο και θα είχε διατακτικό χαρακτήρα και μόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να επιτραπεί μια διαφορετική συμφωνία σε τούτη την περίπτωση, ε, αυτή την περίπτωση μάλλον την εξηγώ ε, ευρέως ε, εις την έκθεση, δεν έχω τώρα χρόνο να την αναλύσω. Ε, πάντως, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή η αρχή δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε αντίθετες ιδέες στη διάρκεια της εξέλιξης του δικαίου και επομένως μπορούμε θεμητά να πούμε ότι έχει χάσει πλέον την ουσία του. Πάντως ε, υπάρχει ε, από τη μία η ιδιωτική ε, de η ιδιωτική ιδιοκτησία από τη μία και το υπόλοιπο δίκαιο από την άλλη. Υπάρχουν στην, στο μόνιμο δικαστήριο Υπάρχουν τμήματα της νομολογίας όπως ας πούμε η υπόθεση Τσίν 1934 ε, ή ε, ας πούμε και μετά από τον ε, πόλεμο για απόφαση του 1952 καθώς επίσης και η έκθεση του πρώτου ειδικού εισηγητή του κυρίου Γκαρσία Αμαδόρ μεταξύ 1956 και 1962, όπως ας πούμε ε, και το δόγμα, όλα αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι τέτοιες ε, ελευθερίες ε, πάντα παρέμειναν εκτός της έννοιας των κεκτημένων δικαιωμάτων. Επίσης καταδεικνύεται ότι δεν έχουν ανεξάρτητη, ανεξάρτητη υπόσταση από τα δικαιώματα και από τα ε, κείμενα και από τις συμβάσεις ε, βάσει των οποίων έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, οι επιχειρηματικές ε, ελευθερίες δεν μπορούν να ισχύουν εάν λήξουν οι συμβάσεις βάσει των οποίων έχουν δημιουργηθεί. Τρίτον, η δυνατότητα διεθνής ε, ε, ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συμπέρασμά μου είναι ότι δεν ε, έχει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν αρνηθεί τα κεκτημένα δικαιώματα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής, της, του Ηνωμένου Βασιλείου όταν αυτό αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, Εάν δεν έχει υπάρξει παράνομη πράξη, δεν υπάρχει ε, ε, και ευθύνη. Η ευθύνη προκύπτει ε, μετά από την διάπραξη παράνομης πράξης. Εδώ δεν έχουμε παρανομία ούτε από πλευράς ε, του Ηνωμένου Βασιλείου που φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε παράνομη πράξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η οποία ε, δεν εξακολουθεί να παρέχει κεκτημένα δικαιώματα στους πολίτες της χώρας η οποία αποσύρεται. Δεύτερον, εάν δεν υπάρχει ε, ε, συγκεκριμένο δίκαιο το οποίο παραβιάζεται, δεν μπορεί να υπάρχει και ευθύνη. Ε, η νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου επ' αυτού είναι σαφής και αναφέρει ότι η οποιαδήποτε ζημία οικονομικού χαρακτήρα, η οποία δεν προκύπτει από οποιαδήποτε παράνομη πράξη από πλευράς των κρατών, δεν μπορεί να εγείρει ε, αξίωση αποζημίωσης. Ε, αυτό άλλωστε ε, κατεδείχθηκε στην απόφαση Ακού Γκιάλο Σάντο. Δεν έχουμε λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση παράνομες πράξεις οι οποίες να εγείρουν αξιώσεις ή ευθύνες. Επόμενο σημείο είναι γεγονός ότι το άρθρο 71β της Συνθήκης της ε, Βιέννης ε, του 69 επί του δικαίου των, συμβάσεων ε, αναφέρει ότι οι χώρες δεν μπορούν να θεωρηθούν υπέτειες για οποιαδήποτε ζημία προκύψει σε περίπτωση που πάψει να ισχύει μια σύμβαση. Ε, αυτό είναι ε, σαφές και από την ερμηνευτική σημείωση ε, της ε, Επιτροπής Ερμηνείας ε, της Σύμβασης και εκεί αναφέρεται σαφώς ότι αναφερόμαστε εδώ σε δικαιώματα των κρατών και όχι των ιδιωτών. Αναφέρει δε η ερμηνευτική σημείωση ότι αναφερόμαστε αποκλειστικά σε δικαιώματα των κρατών και όχι σε δίκαια των μεμονωμένων ατόμων. Ο Σερ Χάμφρι ε, το ίδιο, ο οποίος είναι Βρετανός ε, εισηγητής, ε, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα. Ο ο Λεωφισμόρης και άλλοι. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας σε, αυτήν, σε αυτό το σημείο εν ώψη ενδεχόμενου διαλόγου γιατί έχουν, έχουν αρχίσει αμφίσιμες εμπειρίες, ε, συγγνώμη, ερμηνείες από πλευράς ε, της ε, Βρετανίας. Είναι γεγονός ότι από τη μία πλευρά υπάρχουν τα κεκτημένα δικαιώματα και από την άλλη πλευρά στην 4η ε, Μαρτίου του 2007 2017 ε, η Βουλή των Λόρδων ε, ενέκρινε ε, έκθεση για, την, για τον προϋπολογισμό όσον αφορά τα ρέστα λιγκητέ, τα χρησιμοποιητά αποθεματικά και εκεί αναφέρουν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 91α ή η η εληψη αυτού ε, ε, προσπαθούν να μην ε, εφαρμόσουν το άρθρο 71β έτσι ώστε να αποφύγουν αυτήν την αποσύνδεση του ευρωπαϊκού δικαίου από το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό οι διαπραγματευτές μας να βάλουν όλα τα ζητήματα και να τα αντιμετωπίσουν από κοινού έτσι ώστε να μην προκύψουν δυσαναλογίες και ελλείψεις ισορροπίας. Επόμενο σημείο, η ε, απόσυρση της ε, Γρυλανδίας ε, δεν έχει την ίδια φύση και δεν αποτελεί αντίστοιχο παράδειγμα με την ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά αυτό το οποίο παραμένει εκτός του πεδίου ε, εφαρμογής ε, αφορούσε μονάχα ένα τμήμα ε, του εδάφους της Δανίας και επομένως υπήρξε μία μικρή αλλαγή όσον αφορά τα εδαφικά. Και όπως είπε και η Κομισιόν, η απόσυρση αυτή αφορούσε μονάχα ένα πολύ μικρό αριθμό ατόμων και επομένως δεν είναι συγκρίσιμο με την παρούσα κατάσταση, όμως μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να προβλέψει μία μία μεταβατική περίοδο έτσι ώστε να καλυφθούν τα δικαιώματα αυτών των πολιτών. Φτάνω στο τελευταίο μου σημείο, έκτο και τελευταίο, έστω και αν δεν υπάρχουν και εκτιμένα δικαιώματα τα οποία να μπορούν να παραμείνουν αυτούσια μετά την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου, παρόλα αυτά λέω ε, και σε περίπτωση που δεν ε, συμφωνηθεί μια γενικότερη συμφωνία που να τα περιλαμβάνουν αυτά τα κεκτημένα δικαιώματα, Παρόλα αυτά λέω, τίποτα δεν εμποδίζει ε, τα ε, εθνικά κράτη να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις ε, και διατάξεις για μια συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο με τρόπον ώστε τα συγκεκριμένα άτομα να διέπονται για μια συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο ακόμη από τα ίδια δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό στην επερχόμενη διαπραγμάτευση το περιεχόμενο της οποίας θα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, να εφαρμοστούν οι αρχές ε, της αναλογικότητας ε, ε, και της μη διακριτικής μεταχείρισης για λόγους υπηκότητας και επομένως να μπορέσουν οι πολίτες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου να απολαμβάνουν αυτών των δικαιωμάτων. Υπάρχουν θέματα τα οποία εκ πρώτης όψεως εμφανίζονται ως πολύ απλά. Ένα απλό ζήτημα στο οποίο θα επιμείνει ο συνάδελφος ε, ε, καθηγητής κύριος ε, Γκαρίδο είναι ότι ίσως είναι καλύτερα να υπάρξει έστω μία συμφωνία παρά καθόλου συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά Αντώνιο Φερνάντο Τομάς. Θα δώσω τώρα στο λόγο στον κύριο Διέγκο Λόπες Γκαρίδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ντανούτα Χούμπνερ, αξιότιμοι βουλευτές και αξιότιμο ακροατήριο. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην Επιτροπή ΑΦΚΟ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας ευχαριστώ για την ανάθεση που μας ε, κάνατε να εργαστούμε επί του λεγόμενου Brexit και της ε, επιπτώσεις που μπορεί το Brexit να έχει στους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την νομική υπηρεσία, τον Μιγγέλ Τέλ και τον κύριο Ιωάννη Παπαγεωργίου που μας βοήθησαν που μας βοήθησαν, λέω, ε, και μας καθοδήγησαν στη διάρκεια της ε, διαδικασίας. Ο προκαθηγητής Τομάς αναφέρθηκε στην περίπτωση του διεθνούς δικαίου. Εγώ όμως θα αναφερθώ περισσότερο ε, υπό τη σκοπιά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συνταγματικού δικαίου. να μην ε, λησμονούμε τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη House of Commons τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, εκθέσεις ε, του House of Lords, τις δηλώσεις της Βρετανικής κυβέρνησης, όλα αυτά λοιπόν που συνέβησαν το τελευταίο, το τελευταίο διάστημα. Εξ αρχής, θέλω να πω ότι κατά την άποψή μας τα δικαιώματα των πολιτών, ανδρών και γυναικών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των πολιτών της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, η αντιμετώπιση, λέω, θα πρέπει, αυτών των δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελέσει την πραγματική προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων που ξεκινούν ή θα ξεκινήσουν ανάμεσα από τη στιγμή που η κυβέρνηση της κυρίας Τερέσα Μέη θα καταθέσει σχετικό αίτημα ε, σχετικά με το άρθρο 50 της Εθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία απόσυσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, είναι προτεραιότητα, υπάρχουν βεβαίως και κάποια εκκρεμώντα οικονομικά ζητήματα. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε ότι η ύψιστη προτεραιότητα ε, θα πρέπει να είναι ακριβώς να αντιμετωπιστούν τα δικαιώματα των πολιτών. Τι θα γίνει δηλαδή με αυτούς τους ανθρώπους ε, οι οποίοι είτε ε, είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή υπήκοη μίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή Βρετανοί οι οποίοι ζουν σε μία από τις υπόλοιπες 27 χώρες. Ποια θα είναι η κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι περισσότερα από 3 εκατομμύρια οι ξένοι υπήκοοι οι οποίοι ζουν ε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρέχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 900.000 ε, είναι Πολωνοί υπήκοοι. Και περίπου 1 εκατομμύριο πάνω κάτω Βρετανοί ζουν εκτός της Βρετανικής επικρατείας σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στη δε χώρα μου την Ισπανία. Έχουμε περίπου 300.000 Βρετανούς υπηκόους. Είμαστε η πρώτη ε, ε, χώρα, δηλαδή έχουμε τους περισσότερους Βρετανούς υπηκόους σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει, εξ αρχής λέω να πω, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την ε, συμφωνία ε, που θα επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με, την, με το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει τέτοια συμφωνία μέσα στα δύο χρόνια που προβλέπει άλλωστε το άρθρο που ανέφερα προηγουμένως. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και λόγω αυτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πλήρως θα εμπλακεί σε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση του λεγόμενου, του αποκαλούμενου Brexit. Εγώ θα αναφερθώ σε 7 σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά και πρέπει να αναφερθούν. Πρώτον, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ε, στο πνεύμα των ε, Ευρωπαίων πολιτών, κυρίως ε, δηλαδή και τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν αλλού. Ε, πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο αναφέρεται σαφώ ε, στην έκθεση του House of Commons ε, της Βουλής των Κοινοτήτων τη 5 η Μαρτίου, πριν από μερικέ μέρες δηλαδή και όπου ρητά αναφέρεται η ε, μεγάλη αβεβαιότητα ε, των ε, ανθρώπων που δεν ξέρουν τι θα γίνει με τη δουλειά τους, με τη θέση εργασίας τους, με τη σύνταξή τους και που θέλουν όσο γίνεται πιο γρήγορα να δουν τι θα συμβεί και ποια θα είναι η τύχη τους. Τα άτομα αυτά τα οποία θεωρούν ότι το Brexit θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον τους, θέλουν όσο γίνεται πιο γρήγορα να αντιμετωπιστεί το ερώτημα της κατάστασής τους. Δηλαδή τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους πολίτες μετά από το Brexit. Και αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, ε, στις διαπραγματεύσεις ε, που θρυλείται ότι θα αρχίσουν στις 29 του μηνός Μαρτίου. Δεύτερο. Βεβαίως ο, πυρήνα πυρήνας αυτών των δικαιωμάτων είναι το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ελευθερίας εγκατάστασης. στην Οδηγία 2004 38 που είναι θεμελιώδου σημασίας αναφέρεται μια σειρά ιδιαιτέρως σημαντικών δικαιωμάτων που έχουν οι πολίτες της Ευρώπης έτσι ώστε να κυκλοφορούν μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εγκαθίστανται σε αυτές. Ε, μετά δε πάροδο 5 ετών να έχουν τη δυνατότητα μονίμου εγκαταστάσεως στις χώρες αυτές. Αυτό αποτελεί τον πυρήνα ε, και για αυτών ζητημάτων και γι' αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε τι θα γίνει με αυτό το δικαίωμα εγκατάστασης και εάν θεωρούμε αν αυτό το δικαίωμα είναι και εκτιμένο ή όχι, ε, το δικαίωμα εγκατάστασης, όπως έλεγε ο συνάδελφός μου, ο καθηγητής Αντώνιο Φερνάνδος ε, Τομάσα, από δική του πλευρά είπε ότι δεν πρόκειται για κεκτημένο δικαίωμα και εμείς από πλευράς του διεθνούς δικαίου ε, λέμε ότι δεν αποτελεί κεκτημένο δικαίωμα γιατί από τη στιγμή που φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο σταματάει η ισχύς του ε, ε, ε κεκτημένου γιατί σταματάει η ισχύς ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται επομένω για κεκτημένο, δεν μπορεί να θεωρηθεί κεκτημένο δικαίωμα. Γι' αυτό άλλωστε, ακριβώ επειδή δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα, είναι σημαντικό στη διαπραγμάτευση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου να συζητηθεί το θέμα και να βρεθεί λύση. Γιατί διαφορετικά θα μείνει σε μία νεφελώδη κατάσταση, σε ένα λίμπο όπω λέμε. αν δεν υπάρξει συμφωνία θα εξαφανιστούν εντό εισαγωγικών τα δικαιώματα αυτά, θα πάψουν να υφίστανται και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξέρουν πλέον ε, ε, πού βρίσκονται ε, και θα συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα, η ατελείωτη, την οποία αισθάνονται αυτή τη στιγμή και οι Βρετανοί που ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι καλή την πίστη εγκαταστάθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρώντας ότι η κατάσταση είναι σαφής και σταθερή και ότι μετά από την ε, ε, παρέλευση πέντε ετών θα μπορέσουν πλέον να αποκτήσουν δικαίωμα μονίμου εγκαταστάσεως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό ανατρέπεται τώρα. Τέταρτο σημείο μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση ή εν πάση περιπτώσει ε, τα δύο, στα δύο επόμενα έτη οπωσδήποτε και απολύτως εφαρμόζεται ε, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης κυκλοφορίας. Εξακολουθεί να ισχύει επομένως το δικαίωμα αυτό μέχρι ότου ε, μέχρι ότου ε, αποσυρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Το άρθρο 50 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπει καμία μεταβατική περίοδο και κανένα μεταβατικό ε, δικαίωμα. Και επομένως από τη στιγμή που ε, ε, υπάρξει η κοινοποίηση από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει του άρθρου 50 για δύο χρόνια, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι στις 29 Μαρτίου κατατεθεί το αίτημα και η κοινοποίηση από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, μέχρι τις 29 Μαρτίου του 2019 δεν θα αλλάξει τίποτα στα δικαιώματα. Επόμενο σημείο τα επαπειλούμενα άτομα, αυτά τα οποία ε, έχουν αβεβαιότητα, που δεν γνωρίζουν τι θα γίνει με τη δουλειά τους, με τη σύνταξή τους, ε, τι θα γίνει με την, τα μέλη της οικογένειάς τους ε, όταν θα αποσυρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι λογικό λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να αποφασίσουν να ξεκινήσουν διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων, να κάνουν επομένως εφέσεις ενώπιον των δικαστηρίων. Διότι ε, ε, ε, και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου και μάλιστα να υπάρξει μια καλή συμφωνία η οποία θα, θα, έχει ένα περιεχόμενο γυτνιάζων, παραπλήσιο μάλλον με το περιεχόμενο των σημερινών σχέσεων. Ε, και άλλωστε και το Κοινοβούλιο ε, στο ψήφισμα του της 22ης Ιουνίου παρελθόντος έτους αυτό ακριβώς ανέφερε ότι η σύσταση που μπορεί να γίνει σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών είναι ότι η κατάσταση μετά το Brexit ε, να μην διαφέρει πολύ από την ισχύουσα κατάσταση έτσι ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα να καλυφθούν οι ανησυχίες και τα δικαιώματα βεβαίως των ε, πολιτών που ζουν, ε, Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή πολιτών Βρετανών που ζουν σε άλλες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενο σημείο. Είπαμε ότι η ε, ε, σύμβαση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό, επομένως, το οποίο διέπει το δικαστήριο του Στρασβούργου θα μπορούσε να εφαρμόσει το άρθρο, ιδιαίτερο στο άρθρο 8 της Σύμβασης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 1 του Πρωτοκόλου Ιδιοκτησίας έτσι ώστε να καλυφθούν δικαιώματα ε, ανθρώπων που θεωρούν ότι έχουν ζημιωθεί, ότι έχουν υποστεί επομένως ε, ζημία λόγω ε, είτε της συμφωνίας είτε της έλλειψης συμφωνίας. Η Σύμβαση λοιπόν Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι μια νομική διάταξη η οποία είναι τελείως διαφορετική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως δίνει δικαιώματα στους Ευρωπαίους Ευρωπαίους πολίτες πολύ λιγότερα από ό,τι ε, παρέχονται στους Ευρωπαίους πολίτες βάσει είτε του άρθρου 20 της Συνθήκης Λειτουργίας είτε των ε, περιεχομένων διατάξεων στην Οδηγία 2004 38. Όμως, μπορεί να, ε, ε, μπορούν να γερθούν αξιώσεις βάσει του άρθρου 8 ε, για τους οικογενειακούς δεσμούς ή βάσει του άρθρου 1 του πρωτοκόλου για τις επαγγελματικές καταστάσεις, συμφωνίες κλπ. Τελευταίο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στην κατάσταση των ε, πολιτών της του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και των υπολείπων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από το Brexit και ως επίδραση, επίπτωση αυτού. Είναι πιθανό, είναι δυνατό μετά την ολοκλήρωση του Brexit οι πολίτες των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν λιγότερα δικαιώματα από ό,τι έχουν τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, ε, και, ε, όμως ε, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν περισσότερα δικαιώματα. διότι μπορεί να υπάρξουν ευεργετικέ εξελίξεις όσον αφορά το δικαίωμα κυκλοφορίας και το δικαίωμα εγκατάστασης ε, και επομένως όλα αυτά ε, θα τα απολαμβάνουν οι ε, πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα Φαντάζομαι ότι το έχει λάβει υπόψη του ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τη στιγμή που θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ευρωπαίοι, οι πολίτες που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπωσδήποτε θα έχουν ε, θα έχουν λιγότερο, ε, λιγότερα δικαιώματα ή θα δουν μία συστολή του δικαιώματος κυκλοφορίας ή εγκατάστασης ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, για τους πολίτες των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξει συστολή των δικαιωμάτων τους. Ε, δηλαδή, από τη μία πλευ... Ε, επομένως, από τη μία πλευρά μπορεί να υπάρχει ε, συστολή δικαιωμάτων μίας χώρας, από την άλλη πλευρά θα έχουμε συστολή δικαιωμάτων σε 27 χώρες. Και αυτό βεβαίως ε, ε είναι είναι οπωσδήποτε πιο σημαντικό. Οι πολίτες της ε, οι πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα έχουν συστολή δικαιωμάτων εγκατάσταση και κυκλοφορία σε μία χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πολίτε του Ηνωμένου Βασιλείου θα δουν τα δικαιώματά του να συστέλλονται σε 27 χώρε. αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και φαντάζομαι το έχει λάβει υπόψη και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. αυτά είναι τα κεντρικά προβλήματα τα οποία μα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όσον ούπο ξεκινήσουν οι ε, ότι Σονούπο θα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δηλαδή, ε, άμα την ενάρξη των διαπραγματεύσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα τα οποία προκαλούν μεγάλη βεβαιότητα στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε τώρα να ξεκινήσουμε το γύρο των απαντήσεων. Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω εγώ. για το κατά πόσο πιστεύετε ότι θα υπάρξει ενδεχομένω ε, αλλαγή σε ό,τι αφορά και τον κίνδυνο των, που αντιμετωπίζουν οι πολίτε που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια α, προοπτική, υπάρχει οποιοδήποτε τέτοιο κίνδυνο οραμών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους καθηγητές που ήρθαν εδώ. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω ε, είναι ότι, και, το λέω συνοπτικά, είναι ότι δεν υπάρχουν και εκτιμένα δικαιώματα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τα δύο από τις δύο παρουσιάσεις γιατί εμείς θεωρούσαμε ότι μπορεί να υπάρχει ένα ισχύον δίκαιο το οποίο μπορεί να ε, ε, διατηρηθεί ε, ακριβώς επειδή αυτά τα δικαιώματα θεωρούνται κεκτημένα. Η απάντηση λοιπόν εδώ είναι αρνητική. Δεν υπάρχουν κεκτημένα δικαιώματα. Δεν υπάρχει ε, η δυνατότητα να παραμείνουν ενισχύει τα κεκτημένα, παλαιά κεκτημένα δικαιώματα εάν δεν υπάρξει συμφωνία ε, και όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα και όσον αφορά τα, τα επαγγελματικά κτλ. Ωραία. Εάν λοιπόν περάσουν δύο χρόνια διαπραγμάτευσης και δεν προκύψει συμφωνία. Τότε αυτόματα όταν περάσουν πλέον ε, τα δύο χρόνια, ε, νομίζω ότι ήδη η κυρία Μέη δήλωσε την απόφασή της ε, ανακοίνωσε την απόφασή της ε, να προχωρήσει στην απόσυρση ακόμα και αν δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Ερώτημα λοιπόν θα έχουν τελειώσει, θα έχουν περάσει τα δύο χρόνια. Δεν θα έχει, ας υποθέσουμε, προκύψει ε, μια νέα συμφωνία. Θα πρέπει ε, οι δύο πλευρές ε, να βρουν κάποιες λύσεις για τους πολίτες τους. Μπορεί να μπούμε δηλαδή σε ένα είδος πολέμου εντός εισαγωγικών. Τι θα μπορούσε να, να συμβεί. Μάιτε Πακαζαούντουα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές που ήταν πάρα πολύ σαφείς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από πλευράς του Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνουμε τώρα που οι πληροφορίες λόγω του διαδικτύου ε, ε, προχωρούν. Είχαμε την ε, εντύπωση ότι δεν υπάρχουν και πολλά προβλήματα αλλά τώρα διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν δικαιώματα πέρα των πολλών άλλων εκατομμυρίων που θα δουν συστολή των δικαιωμάτων τους είτε πρόκειται για δικαίωμα εγκατάστασης είτε δικαίωμα άσκησης ε, επαγγελματικής ε, ε, δραστηριότητας κτλ. Είναι πολλά λοιπόν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Έχουμε λοιπόν την διαπραγμάτευση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά όταν θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, ερωτώ, ε, η η στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να είναι ε, να ε, κάνει μια κακή διαπραγμάτευση, δηλαδή ε, να κάνει μια διαπραγμάτευση η οποία ενδεχομένως να μην είναι πολύ καλή για τους πολίτες τους, με την ελπίδα και με την σκέψη, τη δεύτερη σκέψη, ότι μετά θα κάνει διμερείς συμφωνίες έτσι ώστε να βελτιώσει την κατάσταση αυτή και ε, νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι πολίτες ότι ανοίγει το κουτί της Πανδώρας με αποφάσεις τύπου Brexit. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει κυρία Σπινέλη, του ε, καθηγητέ κυρίου ε, Τομάς και Αγκαρίντο. Ήταν ε, εξαιρετικέ οι παρουσιάσεις που μας έκαναν. Και οι δύο λοιπόν επιβεβαιώνουν με πολύ σωστά επιχειρήματα ε, και μάλιστα βασιζόμενοι ε, και σε ε, εκθέσεις της Βουλής των Κοινοτήτων και ιδιαίτερος δε της Βουλής των Λόρδων που υπήρξε πολύ συγκεκριμένη πάνω στο θέμα αυτό επιβεβαιώνουν λέω ότι το θέμα των κεκτημένων δικαιωμάτων θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το λύσουμε άμεσα δίνοντας και μία συγκεκριμένη εντολή ε, κατά την έννοια αυτή. Δηλαδή η τελική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο ε, θα αποτελέσει προηγούμενο, θα εγγραφεί στην ομολογία. γιατί μας είπατε ότι από τη στιγμή που θα πάυσει η ισχύς της, ε, ε, ε, η της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου θα λήξει και η ισχύς του ευρωπαϊκού δικαίου. Ε, εάν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε, θα μπορούσε εν μέρη ε, να ρυθμιστούν κάποια ζητήματα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, αλλά θα παραμείνει αποσπασματική ε, και, και αυτό βεβαίως με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποφασίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να καταλύσει και την, να αποσύρει την υπογραφή του και από την Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όσον αφορά την ε, ενδιάμεση συμφωνία τη μεταβατική συμφωνία. Οπωσδήποτε ε, θα ε, καλύψει κάποια δικαιώματα στη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Τι θα γίνει όμως μετά, θα υπάρξει μια νέα μεταβατική περίοδος μετά από την απόσυρση. Θα... Γιατί δεν κατάλαβα καλά, θα ισχύσει στην μεταβατική περίοδο το δίκαιο. Ε, ε, Βόρεια Ιρλανδία τώρα, συμφωνία Good Friday. Τι θα γίνει σε σχέση με την εφαρμογή σε, αυτό το, σε αυτή την ε, περιφέρεια ας πούμε και τι θα γίνει και με τη Σκοτία. Γιατί εάν αποσχιστεί η Σκοτία το κάνει ακριβώς για να εξακολουθεί ε, να είναι μέλος, μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στη, υπήρξε μια, μια έκθεση ε, της Βουλής των Λόρδων που ζητούσε σε συγκεκριμένη ε, χρονική περίοδο, τρεις μήνες μετά από την ενεργοποίηση του άρθρου 50. Ε, υπάρχει στα έγγραφα του House of Lords. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση. θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο ακριβώς ε, αυτό το κείμενο της Βουλής των Λόρδων και μια σχετική τροπολογία που ε, υπευλήθη. Λοιπόν, ε, χθες μιλήσαμε για τον Ευρωπαϊκό Δήμο και εγώ πρότεινα ε, ε, εγώ είπα ότι πρέπει να υπάρχει ένα συνταγματικός πατριωτισμός, ένα πάθος των Ευρωπαίων να παραμείνουν μαζί. Ε, μου υπόθηκε ότι αυτή η αντίληψη είναι μάλλον πεπαλαιωμένη, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ε, τη συζήτηση για τα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανοώ ότι όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, το το δίκαιο αυτό είναι πολύ προχωρημένο και τώρα το καταλαβαίνουν πολλοί Άγγλοι μετά από το Brexit γιατί αυτό που έχα, αυτό που θα έχαναν ε, όσον αφορά τα δικαιώματά τους δεν τους το εξήγησαν καλά στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για το δημοψήφισμα. Ευχαριστώ, Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Um, Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους δύο καθηγητές για όσα μας είπαν ότι στην ουσία δηλαδή τα μελλοντικά δικαιώματα των πολιτών δεν είναι εξασφαλισμένα. Ανεξάρτητα από το τι θα συμφωνηθεί, στην, ε, στις μελλοντικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτές οι συμφωνίες είτε πρόκειται για τις μεταβατικές συμφωνίες είτε για τη συμφωνία αποχώρησης του άρθρου 50 θα είναι κρίσιμη σημασία. Το πρώτο ερώτημα που έχω να θέσω είναι σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έρθει σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τα δικαιώματα των ε, πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιους εσωτερικούς κανόνες. Υπό ορισμένε προϋποθέσεις όλοι οι πολίτες της έχουν το δικαίωμα να μεταβούν και να εργαστούν σε άλλες χώρες, σε άλλες, άλλα κράτη-μέλη. Όμως το δικαίωμα υπηκών τρίτων χωρών ε, να εργαστούν σε μια χώρα της Ένωσης, αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Όταν λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάψει να είναι μέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα. Άρα, το δικαίωμα ε, ενός Βρετανού πολίτη να διαμένει και να εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται εθνική αρμοδιότητα της εκάστοτε χώρας. Σε ποιον βαθμό λοιπόν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των ε, πολιτών, των Βρετανών πολιτών. Δεύτερο ερώτημα. Ο καθηγητής Τομάς ε, αναφέρθηκε στην ε, Γρυλανδία. Και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ε, θα έπρεπε να ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο της Γρυλανδίας, να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποχωρήσουν όμως η Αγγλία και η Ουαλία. Πολιτικά και νομικά ε, μου φαίνεται μη ε, ρεαλιστικό κάτι τέτοιο, αλλά ε, ιδίως από την νομική άποψη θα ήταν κάτι τέτοιο εφικτό. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη αναφέρθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει, θα υπάρχει ε, ένα τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου του οποίου η πλειοψηφία ε, ε, μπορούν να παραμείνουν Ευρωπαίοι πολίτες. Και μιλώ για τους κατοίκους της, Βορειας, της Βόρειας Ιρλανδίας. Ακριβώ διότι έχουν το δικαίωμα να λάβουν και την υπηκότητα τη δημοκρατία τη Ιρλανδίας. Ε, μπορούν να απολαμβάνουν οι άνθρωποι αυτοί τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη ακόμη και αν δεν διαμένουν στην, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, που έχετε την ερώτησή μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίε και κύριοι, για το γεγονό ότι ήρθατε να μα μιλήσετε σήμερα το πρωί. Αν δεν σα πειράζει να κάνω μια παρατηρήση πρωτού περάσω στην ερώτησή μου. Το πρώτο θέμα λοιπόν που θα ήθελα να παρατηρήσω ω παρατηρήση είναι ότι πολλά από αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί έχουν να κάνουν με συγκεκριμένε συνθήκες. Πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τα βασικά, τις βασικές αρχές της διαπραγματευτική στρατηγικής. Είτε ριζαμέ, είτε το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν χρειάζεται να αποκαλύψει την διαπραγματευτική τη θέση μέχρι ότου επικαλεστεί το άρθρο 50, το οποίο πλάν θα γίνει σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Πολλά από αυτό που ακούσαμε λοιπόν σήμερα και σε προηγούμενε συναντήσει ενδεχομένω να συμβούν, ενδεχομένω και να μην επαληθευτούν. Καταλαβαίνω φυσικά ότι δεν υπάρχει ε, λόγος να μην κοιτάξουμε και το χειρότερο δυνατό σενάριο και την απειλή, ε, την, οποία, την τιμωρία την οποία ενδεχομένω να υπάρχει ο στοιχείο την οποία και ανέφερε ο κ. Γιούγκερ. Ερωτήσει τώρα. Καταρχά. δεν το είπατε, αλλά θα ήθελα να το λάβετε υπόψη. Το θέμα του άρθρου 9, το άρθρο 9 της συνθήκης, σε ό,τι αφορά την ισότητα και το συγκεκριμένο καθεστώς των κατοίκων. Το υπονοήσατε αυτό με σαφήνεια ότι αυτό αποτελεί πραγματικά πάρα πολύ κακή είδηση για οποιαδήποτε άτομο που δεν κατοικεί στη χώρα του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή στην συνθήκη τη Λισαβόνα προκειμένου να υπάρχει εγγύηση, πραγματική εγγύηση και κατοχήρωση των δικαιωμάτων αυτών, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει το άρθρο 9 στη συνθήκη όπω υφίσταται και να ισχύουν και τα όσα είπατε. Δεύτερη ερώτηση. Για πείτε μα ε, δύο λόγια για την ευρύτερη κατάσταση και το πώ συνδέεται με το Ηνωμένο Βασίλειο και την μεταφορά ε, καθημερινώς ατόμων από το Γιβραλτάρ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αγαπητή συνάδελφοι. Λέει η πρόεδρο. Θα ήθελα τώρα να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Καταλαβαίνω ότι έχουμε πολλά ερωτήματα, αλλά στι 10 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Και μετά θα δώσουμε το λόγο στου καθηγητέ, οι οποίοι θα έχουν το λόγο 10 λεπτά κατά κεφαλήν. Αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι. Ποιο θα λέει να πάρει το λόγο. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα απαντήσω στις ε, παρατηρήσεις ε, ε, και ερωτήσεις των βουλευτών. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με τις παρατηρήσεις του κυρίου Αουρέγγινα, να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, ε, ε, τα δύο χρόνια είναι ε, μέση περίοδος και το άρθρο 50 αναφέρει ότι θα μπορούσε να παραταθεί η περίοδος, αυτής, η περίοδος αυτή με ομόφωνη απόφαση. Δεύτερον, σε σχέση με το εάν υπάρξει νέα νομοθεσία. Ναι, όλα αυτά εξαρτώνται από τα διακριτικά δικαιώματα. Όμως, θα ήταν πολύ πιο εύκολο ε, να παραταθούν τα υφιστάμενα ε, δικαιώματα ε, στα πλαίσια της παράτασης. Το νέο νομικό πλαίσιο θα λειτουργήσει, θα καθοριστεί αργότερα όταν θα, έχουν, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Πακάθρο Τουντούα θα ήθελα εδώ να μου επιτρέψετε λογοτεχνική αδεία να σας πω το εξής. Ο τρόπος ε, με τον οποίο να πούμε ε, είτε οι αυτόχθονες φυλές ε, είτε ή στην περίοδο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας στην Ινδία υπήρξε μία δυνατότητα να εξακολουθήσουν τα δικαιώματα των φυλών αυτών θα μπορούσαν να κρατήσουν ένα κοινό ε, μέτωπο, δηλαδή να διατηρηθεί ε, η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης ε, λόγω της εθνικότητας. Αυτό ναι, μπορεί να γίνει υπό την αιγύδα της αρχής της ε, αμοιβαιότητας, ο μου δίνεις και σου δίνω. Σε σχέση με τα ερωτήματα της ε, κυρίας Ασπινέλη Πράγματι, έχω την εντύπωση ότι σε σχέση ε, με την εφαρμοσιμότητα της και δυνατότητα εφαρμογής ε, της ε, συνθήκης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην προκείμενη περίπτωση, νομίζω ότι ωραία ήταν αυτά που είπε η Βουλή των Λόρδων, αλλά δεν εφαρμόζονται όλα πλήρως. Γιατί ξέρετε, για ε, για να μπορεί κανείς να προσφύγει στο ε, δικαστήριο του Στρασβούργου θα πρέπει να έχουν ε, ολοκληρωθεί κάποιες εσωτερικές διαδικασίες. Επίσης οι αποφάσεις δεν είναι δεσμευτικές του Στρασβούργου και τρίτο και σε αυτό συμφωνώ με την κυρία Σπινέλη εάν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διατεθειμένο να, να, να, να φύγει ας πούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως θα αποφασίσει να φύγει και από τη συνθήκη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και επομένως να μην έχουμε ούτε αυτό το πλαίσιο προστασίας. Σε σχέση ε, με ε, μία μεταβατική προσωρινή συμφωνία, ίσως από πρακτικής απόψεως το πιο εύκολο για να λυθεί βραχυπρόθεσμα η κατάσταση θα ήταν ε, μία προσωρινή συμφωνία ε, που θα ενσωματωθεί ε, στην διαπραγμάτευση και που θα καλύπτει τα ισχύοντα δικαιώματα των πολιτών για την ώρα. Τώρα, όσον αφορά διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, θα πρέπει να δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτή η νέα κατάσταση ε, ο κύριος Πέτερ Νόβακ, ας πούμε, ε, είχε κάνει μια εξαίρετη έκθεση στην Επιτροπή ε, λέγοντας, αναφερόμενος σε δικαιώματα τα οποία μπορούν να αντιγραφούν κατά κάποιο τρόπο ή θα μπορούσε να προκύψει μια συμφωνία σου generis σε τελείως διαφορετική από προηγούμενα όσον αφορά Σκοτία και Βόρεια Ιρλανδία. Νομίζω ότι η θέση μου ε, και ως ε, καθηγητού του Διεθνούς Δικαίου αλλά και ως ε, Ισπανός η θέση μου μας είναι σαφής. Βόρεια Ιρλανδία και Σκοτία θα πρέπει πρώτα να αποσχιστούν από το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά ε, να κάνουν οτιδήποτε. Δεν μπορεί να, κάνουν, να δημιουργήσουν ένα είδος γέφυρας, πασαρέλας ε, ε, που να δώσουν την δυνατότητα η Βόρεια Ιρλανδία ή η Σκοτία να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι. Όσον αφορά την τροπολογία της ε, Βουλής των Λόρδων σε σχέση με το κείμενο της απόφαση για την απόσυρση, ξέρετε ότι έκαναν δύο τροποποιητικέ προτάσεις. Ε, η μία αναφέρει ότι όλα θα πρέπει να περάσουν από το Κοινοβούλιο, πολύ λογικό αυτό, ε, είτε αν υπάρξει είτε αν δεν υπάρξει συμφωνία ε, απόσυρσης, αλλά δεν πέρασε. Ε, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Στην πρώτη τροπολογία, η οποία είχε τις καλύτερες προθέσεις από πλευράς των ε, Λόδων, που επίσης δεν πέρασε στην Βουλή των Κοινοτήτων, η τροπολογία έλεγε η εξή ε, και σας το λέω έτσι περιληπτικά, ότι εντός τριών μηνών η αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να διασφαλίζουν ε, στους πολίτες της ΕΟΧ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ιδίους, ε, καθώς επίσης και στα μέλη της ε, οικογένειας που διαμένουν νομίμως στο Ηνωμένο Βασίλειο τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πρέπει, λέει, να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο σε περίπτωση εργασίας και σε περίπτωση εγκατάστασης να παραμείνουν τα δικαιώματα και για το μέλλον. Εγώ βλέπω εδώ δύο προβλήματα σε αυτό το κείμενο, το οποίο ευτυχώς ε, δεν έγινε δεκτό. Ε, πρώτον, η θέση σε ισχύ, δηλαδή η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να παράγεται δικαίωμα ε, θα μπορούσε να είναι η 29η Μαρτίου. Ωραία. Αλλά τι θα γίνει με τα δικαιώματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν οι πολίτες από την ε, ε, αρχή της ενοποίησης μέχρι την αρχή της ε, και της θέσης ισχύς σε συμφωνία. Επίσης, εδώ μιλάμε για μία πράξη η οποία, θα, η οποία αντιτίθεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ε, ότι εξακολουθούν να υφίστανται δικαιώματα των ε, πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν σε άλλες χώρες ε, και των πολιτών άλλων χωρών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και επομένως εάν ακολουθήσουμε, ε, εάν αυτό το κείμενο μάλλον ε, ε, εγκριθεί, τότε σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το εσωτερικό Βρετανικό Δίκαιο δεν έχουν δικαίωμα. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Κόρμπιτ. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιτύχει συμφωνία επί όλων των σημείων με, την, με το Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει να το κάνει Μάλλον όχι, λέτε τι θα γίνει ε, με τους πολίτες τρίτων χωρών. Κοιτάξτε, πρέπει να ξεχωρίσουμε εάν αυτή η τρίτη χώρα έχει ειδική συμφωνία ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε συμφωνία ε, σύνδεσης ή συμφωνία συνεργασίας και επομένως εάν οι πολίτες της χώρας αυτής χαίρουν κάποιων ειδικών δικαιωμάτων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Στο σημείο 70 του πρώτου τμήματος ε, της ε, έκθεσής μου το αναφέρω αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα εξακολουθήσει να παραμείνει ίδια σε σχέση με την ε, τρίτη χώρα, αλλά ε, δεν θα έχει την ίδια κατάσταση το Ηνωμένο Βασίλειο. Οποιοδήποτε δικαίωμα πρέπει να, να διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να το διασφαλίσει εντός της επικρατείας των κρατών μελών που εξακολουθούν να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως θα πρέπει να προκύψει μια νέα συμφωνία με αυτή την τρίτη χώρα από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θα πρέπει ε, επομένως να δούμε τα στοιχεία αυτά σε σχέση με, τον, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από την απόσυρση. Όσον αφορά ε, την Ιρλανδία, την ε, Σκοτία, ε, η απάντησή μου είναι σαφώς αρνητική. Δεν υπάρχει σχέση. Η Ιρλανδία είναι τμήμα μιας χώρας μέλους και επομένως η έξοδος της Ιρλανδίας μπορεί να είχε μια αλλαγή της της χωρικής εφαρμογής, εδαφικής εφαρμογής του δικαίου, αλλά δεν απέτησε οποιαδήποτε ε, άλλη ε, τροποποίηση του δικαίου ή οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση ε, των κρατών μελών. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να εξομοιωθούν οι δύο καταστάσεις. Υπάρχουν και για πολλούς λόγους μάλιστα. Οι κάτοικοι της ε, ε, Γρυλανδίας, ε, οι οποίοι ψήφισαν, ας πούμε, στο δημοψήφισμα ήταν περίπου 32.000, ενώ ενώ, ε, α, επίσης ε, υπάρχει ένα ε, έγγραφο, το 1 κάθετος 83, το, είναι έγγραφο της Επιτροπής που αναφέρει ότι ήταν εξαιρετικά μικρός ο αριθμός των ατόμων που που ε, εφήγησαν από την κατάσταση, από την απόσταση της ε, Γρυλανδίας. Ε, το ζήτημα εδώ είναι τελείως διαφορετικό. 11, χρόνια μόνο η Γρυλανδία υφίστατο ας πούμε το κοινοτικό δίκαιο και επομένως δεν είχαν, δεν είχαν δικαιώματα συνταξιοδοτικά οι κάτοικοι της ε, Γρυλανδίας. Όμως είχαν ε, κεκτημένα δικαιώματα. Χρησιμοποίησε η Κομισιόν εσφαλμένα κατά την άποψή μου την έννοια των κεκτημένων δικαιωμάτων με την έννοια δηλαδή ότι ε, είχαν κάποιες θεμητές προσδοκίες όσον αφορά την συμμετοχή της Γρυλανδίας. Η Κομισιόν η Κομισιόν στην ε, ε, συμφωνία τροποποίησης ε, της συμφωνίας η Κομισιόν λέω αναφέρθηκε σε κεκτημένα δικαιώματα και επομένως αυτό οδήγησε στην προστασία αυτών των ανθρώπων. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει όμως πρότυπο για την προκείμενη κατάσταση Γιατί εάν πούμε ότι ε, η συμφωνία της, ε, ε, ότι η διαπραγμάτευση, η προσωρινή συμφωνία ή η μελλοντική συμφωνία δεν μπορεί να προβλέψουμε ότι θα σέβεται και θα εξακολουθεί τα κεκτημένα δικαιώματα. Τέλος. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Τζέιμς. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα αποκαλύψει τη θέση της η κυρία Μέη θα είναι καλό γιατί ε, θα ε, ξέρουμε ε, τι ακριβώς επιθυμεί και που θέλει να βασιστεί. Μακάρι να ξεκαθαρίσει γρήγορα τα μελλοντικά της σχέδια όσον αφορά το άρθρο 9 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορώ να σας πω ότι το άρθρο 9 λέει ότι ε, θα γίνει σεβαστή η αρχή ε, ε, της ισότητας των πολιτών. Αλλά αν συνεχίσετε την ανάγνωση λέει ότι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοείται οποιοδήποτε πολίτης έχει την υπηκότητα μιας χώρας μέλους. Επομένως, εάν πάυσει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ηνωμένο Βασίλειο, επομένως δεν χαίρουν πλέον αυτής της ιδιότητας οι πολίτες του όσον αφορά το Γιβραλτάρ. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ε, ζήτημα το οποίο προκύπτει διαρκώς ε, ε, στις σχέσεις και στις συζητήσεις μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Ξέρετε πάντως ότι το Γιβραλτάρ ε, ε, είναι λίγο αναχρονιστικό, αλλά παρόλα αυτά ε, πρόκειται για, ένα, για μια επικράτεια η οποία βρίσκεται σε μεταπικιακή κατάσταση. Εδώ δεν αναφερόμαστε στην, στο δικαίωμα εγκατάστασης ή οτιδήποτε. Δεν νομίζω ότι ε, η Ισπανική κυβέρνηση προτίθεται να επιστρέψει στο ε, παρελθόν. Ε, η θέση της Ισπανίας, έτσι όπως αναφέρθηκε και ενώπιον ε, της τετάρτης ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, παραμένει ε, ανοιχτή, δηλαδή παραμένει η δυνατότητα της διπλής υπηκότητας της Ισπανικής Βρετανικής, μιας ειδικής φορολογικής κατάστασης και γενικότερα ενός ειδικού καθεστώτος που δεν μου φαίνεται να προκαλεί οποιοδήποτε πρόβλημα προς ώρας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Γκαρίδο. Ο κύριος Διέγκο Λόπες Γκαρίδο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από τις παρεμβάσεις ε, και τις ερωτήσεις προκύπτει ένας κοινό τόπος ε, που επικεντρώνεται στις συμφωνίες, τις ακόλουθες συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Σύμφωνα με το άρθρο 50 υπάρχει μια αρχική συμφωνία η οποία θα έχει διάρκεια διετή που θα ξεκινήσει από τις 29 Μαρτίου αν υποθέσουμε ότι όντως ε, <coughs> ισχύσει η κοινοποίηση της διαδικασίας. Ε, επομένως, στη διάρκεια αυτών των δύο ετών, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, παραμένει, παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Εάν εντός των δύο ετών δεν προκύψει συμφωνία, αυτόματα θα αποσυρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός και αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίσει παράταση αυτής της περίοδου. Αυτό που λέμε εμείς ε, είναι ότι σε αυτήν την αρχική ε, απόφαση απόσυρσης το Ηνωμένο Βασίλειο ως πρώτο ερώτημα ως πρώτο ζήτημα και πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα των δικαιωμάτων των πολιτών, γιατί είναι πολλά εκατομμύρια πολιτών που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά μεγάλη αμβεβαιότητα για το μέλλον τους. Ε, ε, είτε ζουν στο, ε, ως πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε πολίτε του Ηνωμένου Βασιλείου σε άλλε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την ίδια αβεβαιότητα. Δεν μπορούν να περιμένουν ε, δύο χρόνια για να δουν τι θα του συμβεί στο μέλλον, να δουν ποιο θα είναι το μέλλον του. Επομένω, στην αρχική συμφωνία, την αναφερόμενη στο άρθρο 50, θα πρέπει εξ αρχή να γίνει λόγο και να αντιμετωπιστούν τα ε, δικαιώματα των πολιτών. Αυτό είναι κατεπήγον κατά την άποψή μου. Αυτό όσον αφορά την αρχική συμφωνία. Από τη στιγμή που υπάρξει συμφωνία. Και βεβαίως μέχρι τότε νομικά ε, είναι όλοι έχουν ε, την ε, ίδια αντιμετώπιση γιατί εξακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι περάσουν τα δύο χρόνια και δεν έχουμε συμφωνία, τότε αυτόματα πάβει το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή τη στιγμή, μετά την πάροδο δηλαδή των δύο χρόνων, ενδεχομένως να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια μεταβατική συμφωνία πριν από την παρέλευση των δύο ετών. Με, αφού παρέλθουν τα δύο έτη, ενδεχομένως προκύψει μια μεταβατική συμφωνία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα πιο σοβαρά θέματα μέχρι ότου ε, φτάσουμε σε μία τρίτη συμφωνία που θα είναι η τελική συμφωνία η οποία θα αποτελέσει το τελικό πλαίσιο ε, των σχέσεων που θα διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο έτσι όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 και το οποίο θα αποτελέσει νέα ε, συνθήκη. Και επομένως τότε πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πλέον τρίτη χώρα και θα μπορεί να κάνει επιμέρους συμφωνίες. Άρα έχουμε τρία είδη κειμένων, ε, τρία είδη συμφωνίας. Ε, το πρώτο, το οποίο ε, θα είναι μέχρι τα δύο χρόνια και που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα λόγω της αβεβαιότητας προκαλεί. Δεύτερο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η απόσυρση να υπάρξει ενδεχομένως μια μεταβατική συμφωνία έτσι ώστε να ε, λυθούν εκρεμή επίγοντα ζητήματα και μετά θα έχουμε την τρίτη τελική συμφωνία που θα διέπει τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα είναι βεβαίως και μια συμφωνία ευρυτάτη και η οποία ε, θα αναφέρεται σε όλα τα επιμέρους ε, σημεία. Αυτή είναι η διαδρομή των συμφωνιών ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Εξ αυτού, γιατί μέχρι τώρα απαντούσα σε αυτά που είπε ο κύριος Χαουρέγγι. Όσον αφορά την ε, κυρία Τουντούα, ναι, μπορεί να υπάρξει στρατηγική από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου να, ε, ε, ε να διαβουλευθεί, να, να κάνει διμερείς συμφωνίες με κάθε μία από τις χώρες και να μην κάνει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είναι σαφής η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δηλαδή θα πρέπει η συμφωνία να είναι μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, και Ηνωμένου Βασιλείου εν το συνόλο της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και όχι με τις μεμονωμένες χώρες. Και η πρώτη συμφωνία και η δεύτερη και η τωρινή και αυτή η μετέπειτα όταν δεν θα είναι μέλος πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να είναι σαφείς, αναλυτικές και λεπτομερείς έτσι ώστε να μην αφήνουν περιθώριο για διμερείς συμφωνίες. και άλλωστε και το άρθρο 218 της συνθήκης αναφέρει ότι το Συμβούλιο θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές ε, της διαπραγμάτευσης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ε, που θα εγκριθούν από το Συμβούλιο οπωσδήποτε τις επόμενες μέρες είναι υψή τη σημασίας, διότι θα πρέπει να προσανατολίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στις σωστές ε, κατευθύνσεις. Ε, προς τις κατευθύνσεις τις οποίες εμείς αναφέρουμε στην έκθεση. Ε, αυτές έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αυτές είναι ε, αυτές οι οποίες θα αποφύγουν τον κίνδυνο των διμερών πούμε συμφωνιών και της διμερούς αντιμετώπισης σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Σπινέλη. όντω ε, μπορεί να έχει ισχύ και να ισχύσει και να εφαρμόζεται η συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι ε, δεν θα αποσυρθεί από αυτήν το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, όσον αφορά την ερώτηση που κάνατε για τη μεταβατική συμφωνία, νομίζω ότι ήδη σας κάλυψα και απήντησα, δηλαδή είπα ότι αυτή τη στιγμή και μέχρι δύο χρόνια δεν αλλάζει τίποτα, ε, άλλωστε το άρθρο 50 δεν ε, επιτρέπει μεταβατική συμφωνία, ε, ε, δίνει τη δυνατότητα μόνο για μία συμφωνία, όχι δύο. Από την παρέλευση των δύο ετών και πέρα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ενδεχόμενη μεταβατική συμφωνία. Όσον αφορά δε την πρόταση ε, του House of Lords και House of Commons, Πρόκειται όντως για πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα και πολύ επικοδομητικά. Νομίζω ότι η θέση της Βουλής των Λόρδων και της Βουλής των Κοινοτήτων στο κείμενο που ονομάζεται Governments Negotiation Objectives διαπραγματευτική στόχη της κυβέρνησης εν ώψη ε, της ε, ε, συμφωνίας, της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι είναι ανάγνωσμα εξαιρετικά ενδιαφέρον και συμφωνώ με την κυρία Σπινέλη ότι δηλαδή πολλά χάνουν και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι πολίτες του φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θα χάσουν δικαιώματα σε 27 χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωση ε, που πρόκειται για μια θεαματικά ευρεία γκάμα, ένα ε, εξαιρετικά ευρύ φάσμα ε, δικαιωμάτων όσον αφορά την εγκατάσταση, όσον αφορά την εργασία, όσον αφορά την διαμονή, όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και επομένως όλα αυτά τα χάνουν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου με την απόσυρση τη χώρα από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει όμως, για, για μας που δεν θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θα εξακολουθήσουμε να απολαμβάνουμε τα δικαιώματα αυτά σε 27 χώρες και αυτό ήδη είναι θετικό. Τέλος, αυτά που είπε ο κύριος Ρίσορ Κόρμπεντε, νομίζω ότι πολύ καλά τα είπε ο συνάδελφος Αντώνιο Φερνάντες Τομάς. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως μπορεί να διατηρήσει κάποια δικαιώματα, μπορεί να το κάνει, οι σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διέπονται ε, από μία αρχή, ε, η οποία είναι η αρχή της ε, αμοιβαιότητας και την οποία άκουσα και από, την, από τους ίδιους τους Βρετανούς. τώρα, ναι, αναφέρεται η κυρία Τζέιμς σε συγκυρίες, μα ίσα ίσα εμείς δεν θέλουμε συγκυριακή αντιμετώπιση, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρξει συγκυριακή αντιμετώπιση έτσι ώστε να αρθούν οι αβεβαιότητες, η αίσθηση κινδύνου, ε, που είναι μια αίσθηση που την έχουν πλέον εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, μάλλον εκατομμύρια ε, πολίτε που δεν ξέρουν τι θα γίνει με την οικογένειά του, τα μέλη τη οικογένειά του, με τη δουλειά του, με τη σύνταξή του ε, τα δικαιώματά του, τι θα γίνει με του φοιτητέ που ζουν αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο και που θεωρούμε ότι αυτή η αβεβαιότητα είναι κάτι εξαιρετικά αρνητικό. Το είπα και στην αρχική μου εισήγηση και γι' αυτό ακριβώς είπα ότι θα πρέπει είναι κάτι το οποίο θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί και να λυθεί και αυτό νομίζω ότι είναι και το κεντρικό μήνυμα το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε μέσω ε, του, ε, της έκθεσής μας και ε, ο συνάδελφος Τομάς και εγώ ο ίδιος. να υπάρξει μια καλή συμφωνία για αυτούς που ήδη σήμερα απολαμβάνουν ακριβώς των δικαιωμάτων του, του να είναι πολίτες της Ευρώπης, 4 εκατομμύρια στο σύνολο, 3 εκατομμύρια ξένοι στο ΕΒ, Βασίλειο, 1 εκατομμύριο ε, Βρετανοί σε, τρίτες, ε, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτούς η καλύτερη δυνατή συμφωνία, αλλά και η καλύτερη δυνατή συμφωνία όχι μόνο για αυτούς ε, που ζουν ήδη, αλλά και για το μέλλον γενικότερα. Για αυτούς που ε, είτε θα θελήσουν κάποια στιγμή να ζήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε και για τους Βρετανούς που θα θελήσουν κάποια στιγμή να φύγουν από την ε, ε, χώρα τους, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις η βέλτιστη δυνατή συμφωνία είναι η μόνη καλή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και τους δύο καθηγητές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως για τις παρεμβάσεις σας αυτές και έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή θα γίνει η επίκληση των άρθρων και θα ξεκινήσουν οι πραγματεύσει, Θα επανέλθουμε σε κάποια τα θέματα τα οποία ακούσαμε σήμερα. Πολλά εκκρεμή ζητήματα, κυρίω το θέμα τη ε, δικαιοδοσία για τα διάφορα ζητήματα, για τι διάφορε συμφωνίε. Ε. Άρα πολλά από αυτά τα θέματα τα οποία ακούσαμε σήμερα θα χρειαστεί να ξανακοιτάξουμε 100%. Μια ε, αυτή τη στιγμή θα μπούμε πραγματικά στη διαδικασία. Ευχαριστώ και τώρα να πω στου συναδέλφου και πάλι ότι η τελική εκδοχή της έρευνας σε μία εβδομάδα ή ίσως και λίγο παραπάνω να μας διαμοιραστεί από την Γενική Διεύθυνση. Το κλείνουμε λοιπόν το θέμα αυτό και να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Dear colleagues, I would like to start the vote. Να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, συνάδελφοι. It looks like it's, it's not many people, no? Dear colleagues, can we start the vote? Να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, συνάδελφοι. Έχουμε μία ώρα και δέκα λεπτά στη διάθεσή μας. Can we check whether our cards να δούμε κατά πόσο οι κάρτες μας ε, δουλεύουν, αν θέλετε. Δοκιμάστε τις ε, συσκευέ να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Τσεκ. Συνάδελφοι, για ψηφίστε. Γιατί έχουμε και πολλούς συναδέλφους που ακόμα δεν έχουν ψηφίσει. Ένα άτομο μας λείπει. Όχι, εντάξει, 23 ψήφοι. Δύο απόντες. Ξεκινάμε λοιπόν τις ψηφοφορίες και ξεκινάμε με την γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το European Deposit Scheme. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται Deposit Insurance Scheme. Περνάμε στην τροπολογία 2. Α, δεν το ψηφίζουμε. Τροπολογία 2. Την οποία θα τη βρείτε στη δεύτερη σελίδα. Δεύτερη λοιπόν τροπολογία υπέρ κατά. Υπέρ, συγγνώμη. Η τροπολογία 2, παρακαλώ, στη δεύτερη σελίδα, επαναλαμβάνει η Πρόεδρος. Υπέρ. Ξανά. Οι σοσιαλιστές... Οι δύο καλέ. Ε. Dos. Yeah. So who's in favor? Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τρία. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η πέντε Με προφορική τροπολογία. Κανείς δεν είναι κατά της προφορικής τροπολογίας. Ποιος είναι λοιπόν υπέρ της πέντε, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 29 υπέρ. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχο παρακαλώ για την τροπολογία παραθμών 29. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Can you Απορρίπτεται. Μέσο ψηφία 11 και 11. Ή 30 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ και την 31 ηλεκτρονικά. Έναρξη. Εγκρίνεται. Η 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε. Unblock 7 Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Άλλα μου λέει η δεξιά μου και άλλα η αριστερά μου. Άρα θα κάνω το κεφαλιό μου. Υπέρ της τροπολογίες 7 έως 9. Κατά αποχές αγκρίνεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Unblock 12, 15, 16 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνονται. 34 υπέρ κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 34. Έναρξη. Η 34 σε πολλές γλώσσες. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 35 προφορική τροπολογία. Η 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 τώρα. Η 19. Αντιλογικές σκέψεις. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίθηκε με 15 ψήφους υπέρ, 3 κατά, 6 αποχές. Και τώρα περνάμε στα δύσκολα. Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα. Πείτε μου ότι είστε έτοιμοι. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Σεμιβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία. 3. Μάλλον συμβαστική 3. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. I have nobody. Yeah. Σας παρακαλώ να κοιτάξουμε πού βρισκόμαστε. So on compromise three we have... Συμβαστική 3 με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Ψηφίζουμε. We have compromise 3. Συμβαστική 3 με ονομαστική κλίση. Πέρας. And it is rejected. So now we... Απορρίπτεται. Συμβαστική 4, υπέρ. Η συμβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική 6, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική 7, υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 7. Έναρξη ψηφοφορίας. It Εγκρίθηκε με 14 υπέρ 10 κατά. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχέ Και νομίζω ότι εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Ή 48 κάτω-κάτω. Υπέρ. Ή 48 λέω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 11. Εγκρίθηκε. 13. Η συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 14. Συμβαστική 14. 14 παρακαλώ ψηφίζουμε την συμβαστική 14. Πέρας. Εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 59. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 63 και 64. Υπέρ. Ονομαστική κλίση, παρακαλώ. The We have a roll call. Yeah, we have να ξαναξεκινήσουμε παρακαλώ την 63 και 64 ηλεκτρονικά με ονομαστική κλίση. Closed. And it is 16 to 7. εγκρίθηκε 16 πέρα, 7 κατά. Στην 17, στην 70, συγγνώμη, ονομαστικά, με ονομαστική κλίση. Για την 70, ψηφίζουμε. πρέπει να την ψηφίσουμε. Όχι. Excuse me, Chair. It actually for... Πρόεδρε, καταπίπτει. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Η 17. Ξεμιβαστική 17. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 18, συμβαστική 18 υπέρ, κατά. συμβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά αποχές επίσης εγκρίθηκε. 91, η τροπολογία 91 υπέρ, 91 λέω. Υπέρ. Κατά. Α ας ελέγξουμε παρακαλώ την 91. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Παρακαλώ. Κατά. Οι σοσιαλιστές υπέρ. Εγκρίθηκε. 96. 97 υπέρ. Κατά αποχές απορριφθήκε. Ενενήντα εννέα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 99. Υπέρ. Κατά. Όχι ηλεκτρονικά πρέπει να το ελέγξουμε. Πρόεδρε, να σα βοηθήσω λίγο. Νομίζω ότι κάνετε δύσκολη δουλειά γιατί οι συνάδελφοι μπροστά, το ΑΕΛ και το Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες δεν σηκώνουν το χέρι του. Το ξέρω. Και ίσω θα ήθελα να σηκώνουν ε, το χέρι του, μήπω να προχωράμε λίγο πιο γρήγορα κιόλα. Κοιτάξτε, δεν το λέει ο κανονισμό, δυστυχώ, ε, λέει η πρόεδρο, Ελπίζουμε ή πίεση από τους συναδέλφους να δουλέψει. 99 λοιπόν, τροπολογία 99 υπέρ. Κάτα. Ας ελέγξουμε την 99. Εγκρίθηκε 18 υπέρ 6 κατά. 101. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Στην 110 πάμε τώρα. Επόμενη σελίδα. 110 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 115 υπέρ. Κατά. Χρειάζεται έλεγχος εδώ. Για την 115. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 13 υπέρ, 11 κατά. Συμβιβαστική 25. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 26. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 124. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 128. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 128. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκε και πάμε στην 129. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 27 συμβαστική, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 137 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 151 υπέρ, υπέρ, κατά. Κατά αποχές απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά. 152 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε την 152 παρακαλώ. Πέρας. 16 υπέρ, 7 κατά, εγκρίθηκε. 154 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 154 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 160 τώρα. 160 λέω. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 41. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την ε, συμβαστική 41. Έλεγχος. Δύο ψήφοι μας λείπουν. Πέρας. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. So there's a mistake. Two. Now we go to 42. Compromise 42 in favor. Συμβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 45 ονομαστική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 16 υπέρ 8 κατά. 2.59. Επόμενη σελίδα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.62. Υπέρ, κατά. Να σφίσουμε ηλεκτρονικά. Επί της 2.62. Ψηφίστε παρακαλώ. 10 προς 12 απορρίπτεται. Συμβαστική 46 υπέρ, ονομαστική ψηφοφορία εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται 14 προς 9. 47 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 272 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ...271 υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 271 περαση της ψηφοφορίας εγκρίνεται 2.73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.76 υπέρ, κατά, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Vote Πέρασε, εγκρίνεται. 281 υπέρ, κατά, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και για την 281. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίας. Επίσης εγκρίνεται. Συμβαστική 52 υπέρ κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Then we Πέρας. Δύο συνάδελφοι δεν ψήφισαν. Εγκρίνεται. Με 14 υπέρ, 8 κατά. 22 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 282 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 283 υπέρ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά πέρας εγκρίνεται συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές ...285, 286, 2.87 και 2.88 τις ψηφίσουμε από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 2.92 από κοινού με τις 2.93, 94, 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 323 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 342 ε, 324 υπέρ κατά εγκρίνεται 325 να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβαστική 57 υπέρ προφορική τροπολογία ε, διαφωνεί κάποιος με την προφορική τροπολογία όχι άρα την ψηφίζουμε μαζί με την τροπολογία, την προφορική. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην 363, την οποία όμως δυστυχώς δεν μπορώ να βρω. Ε, είναι λάθος. Τι κάνω λοιπόν. Οπότε, όπως ακριβώς είχα πει εξ αρχής, πάμε στην 58. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 369, η οποία έχει αποσυρθεί. Ωραία, 59 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 Υπάρχει προφορική τροπολογία, δεν διαφωνεί κανεί Υπέρ, κατά, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 60 με την προφορική τροπολογία. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται. Πάμε στην 61. Μακριά, μακριά. Υπέρ της 61 να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Φαίνεται σαν να έχει απορριφθεί. Πέρας εγκρίνεται. 62 που είναι στην επόμενη σελίδα. Υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 62. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 63 εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. 64 να μην ψηφιστεί. Πάμε στην 405. Ψηφίζουμε υπέρ κατά ε, οι σοσιαλιστέ ψήφισαν υπέρ. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Η την τροπολογία 305. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 65. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 66. Υπέρ κατά Σοσιαλιστές κατά, οπότε δεν ξέρω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Μάλιστα, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ντροπή μας. 4-16 υπέρ. Υπέρ. 4-16. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 417 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 418 εντάξει. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την ε, τροπολογία 417. Ψηφίστε παρακαλώ. να ξαναψηφίσουμε μάλλον ηλεκτρονικά και για, για την τροπολογία 416. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 416. Εγκρίνεται και αυτή. Εγκρίνονται και οι 416 και οι 417. Πάμε στην 418. Υπέρ, κατά. Ίδια πλειοψηφία. 419. Υπέρ, κατά. Ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία εγκρίνεται. 420. Υπέρ κατά όχι απορρίπτεται 421 ε, υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι και αυτή εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία συμβαστική 57 υπέρ 57 υπέρ 50 67 ε, ε, υπέρ κατά αποχές 68 ε, υπέρ κατά να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά 68 the vote is open ψηφίστε παρακαλώ uh, no, we are on time, so it's, ε, it's 14 to 8, so it's adopted. So now... Εγκρίνεται. 4.28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4.29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4.30. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται με 13 υπέρ, 11 κατά. Συμβαστική 69. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.35. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 448 υπέρ κατά να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 448. Ψηφίστε παρακαλώ. Κάποιος απεργεί και αρνείται να ψηφίσει. Πέρασε. Απορρίπτεται. 450 υπέρ. 450 υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίπτεται με 11 προς 2. Πάμε στη συμβαστική 73. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 455 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ ονομαστική. Δεν, ήθι, δεν, δεν ήθιστε να έχουμε ονομαστικές ψηφοφορίες εδώ στην Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Μάλιστα, 23. Τι λέτε. Και πάμε τώρα στην 76. Όχι, την 76 μόλις την ψηφίσαμε. 77. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 459. Υπέρ κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. 459. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 462. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται λέτε. Να, ξαναψ... να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 462. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 463. Υπέρ. 463 τι λέτε. Έχουμε μια διαφωνία εδώ πάνω. Ωραία, 465. Υπέρ. Rejected. It was rejected, the deletion. So we have to vote. Yes, yes. But no, but we go to the following paragraph. That is new one. Okay. We have to go to new paragraph, so we have to vote amendment for... Θα πάμε σε νέα παράγραφο, οπότε πρέπει να ψηφίσουμε για την τροπολογία 465. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 466. Ναι, πρέπει να τη θέσουμε σε ψηφοφορία, όχι. Ψηφίσαμε. So we have to vote for also, as Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν για την 466 ε, υπέρ κατά. νομίζω ότι εγκρίνεται, γιατί την υποστηρίζουν και οι σοσιαλιστές. Οπότε πάμε στην τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 84. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ε, γιατί διαφωνούν οι σοσιαλιστές. Α, υπερψηφίζεται. Εντάξει, τότε ας πούμε ότι εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία ονομαστική Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ένα μέλος της Επιτροπής δεν έχει ψηφίσει. Παρ' όλα αυτά, κλείνουμε την ψηφοφορία και εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. 20 υπέρ, 2 κατά. Πρόεδρε, μπορώ να σας ζητήσω κάτι πολύ ευγενικά. Υπάρχει λόγος που χρησιμοποιούμε ε, αραβικούς αριθμούς και όχι λατινικούς. Δεν ξέρω ποιος θεώρησε ότι ήταν καλή ιδέα να χρησιμοποιηθούν λατινικοί αριθμοί. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν κάποιος Ιταλός. Μπορούμε να επανέλθουμε στους κανονικούς αριθμούς που ξέρουμε όλοι να διαβάζουμε, γιατί αλλιώς μπερδευόμαστε. Συνάδελφοι, προτού δώσω το λόγο σε εσάς, Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που, που, που το είπες. Παρ' όλα αυτά... Έχουμε ξεχάσει και να διαβάζουμε τους, ε, τους λατινικούς αριθμούς. Οπότε μπορεί και να εξασκούμε και λίγο το μυαλό μα. Έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. <laughs> Εν πάση περιπτώσει, έχουμε χρόνο λίγο. Ε, μην ανησυχείτε, θα σα δώσω το λόγο. Να σα ευχαριστήσω όλου για την ψηφοφορία. Ε, είχαμε κάνει τη συμφωνία ε, ε, ε, ότι θα επανέλθουμε στους αριθμούς του λατινικούς. Εν πάση περιπτώσει, έχεις το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο ήθελα να κάνω σχετικά με τις αραβικές και λατινικές παραδόσεις γύρω από τους αριθμούς. Εγώ θα έλεγα να ε, χρησιμοποιήσουμε λατινικούς αριθμούς, ιδίως αν μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση, γιατί μπορώ να πω ότι τα λατινικά μου άρεσαν πολύ στο σχολείο. Πέραν αυτών, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Τους ευχαριστώ για την υποστήριξή τους. Κάποιοι βέβαια είναι δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα, δεν πειράζει. Ε, εγώ ανακουφίζομαι και χαίρομαι πολύ που ολοκληρώσαμε αυτή την πληροφορία και ότι θα πάει στην ε, Ολομέλεια, γιατί η έκθεση αυτή είναι γεμάτη από προτάσεις για το, προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή και αξίζει να συζητηθεί σε βάθος και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Ρίτσαρτ Κόμπερτ για την ε, ε, συνεργασία του ε, στο πλαίσιο της σύνταξης της δικτύου έκθεσης. Αναγκαστήκαμε να συνεργαστούμε παρότι δεν το θέλαμε κανένας από τους δυο μας να συνεργαστούμε. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τον κύριο Πλάνκοβιτς που δούλεψε πολύ ε, για όλα αυτά, παρότι βρίσκεται τώρα πια στην Κροατία. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε και φυσικά την ευθύνη για τους λατινικούς ε, χαρακτή, για, τα, για τα λατινικά, ε, για τους λατινικούς αριθμούς είναι, την αναλαμβάνω πλήρως εγώ. Δεν ξέρω ποιος επινόησε αυτό το σύστημα ρύθμισης, <laughs> αλλά τι να κάνουμε. Ευχαριστώ ε, πολύ. Ε, τελειώνει η συνεδρίασή μας. Επόμενη συνεδρίαση